Χαίρομαι για την παρουσία του προεδρίου του Βόρειο Σκανδιναμικού Συμβουλίου με την παρουσία της κυρίας Ούνουρ Μπρακράντα Οντοστήρ από την Ιλλανδία και του Μπιλ στην Ουσέν από τα νησιά Φαρόε που είναι στην, στο, στα θεωρία των επισήμων. Πολλοί συναδελφοί μα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με του συναδέλφου από τα νησιά Φαρόα και την Ισλανδία και να συζητήσουν πολλά θέματα, ιδίω θέματα αλληλεία στον Αρκτικό ωκεανό. Χαιρόμαστε που μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο μαζί του. Και θέλω και πάλι να του ευχαριστήσω για την επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση ΕΕΛΑ, κανόνε για τη συμμετοχή στον ορίζοντα 2020. Καταρχήν ψηφίσουμε